Ευρώπη των Ελευθεριών και της Δημοκρατίας. Από τους σοσιαλδημοκράτες έχω ένα αίτημα η κυρία Φραντσέσκα Μπαρατσού να διοριστεί ως μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού διορίζεται. Υπάρχουν κάποιες ενστάσεις? Δεν υπάρχουν. Έτσι αυτός ο διορισμός ε, κυρώνεται. Η ακόλουθη γραπτή δήλωση έχει υπογραφεί από Ευρωπαϊκή